Ε, ε, λοιπόν, να σας εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι προεδρεύω βάσει του άρθρου 213 και μόνο αντιπρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων ήμουνα και θα παραμείνω εδώ μέχρι να ορίσουμε τον νέο μας πρόεδρο. Λοιπόν, η συνάντησή μας σήμερα προβλέπεται για να συγκροτηθεί σε σώμα η Επιτροπή μας και να εκλέξει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους βάσει του άρθρου 213. Τώρα προβαίνουμε στην ψηφοφορία του Προέδρου. Όπως γνωρίζουμε, ε, τα αναπληρωτικά μέλη τα οποία συμμετέχουν σήμερα θα πρέπει να καθίσουν στις θέσεις των μελών που αντικαθιστούν και να το πούν αυτό στη γραμματεία. Θα σας διαβάσω τώρα ποιος αντικαθιστά πλήρη μέλη για το έλικα. Μέντα αντικαθιστά την κυρία Χουμπνέρ. Για τους σοσιαλιστές δεν μας έχει ανακοινωθεί η αντικατάσταση. Για την ανέωση της Ευρώπης Κραβάτσεφ αντικαθιστά την κυρία Σαστέλ και συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά τα ονόματα, λέει ο πρόεδρος. Για το IND, ε, κύριε Ντονάτο, αντικαθιστά, κύριο Ζάνε, για το ECR. Η Τζέσικα Στέγκρου το αντικαθιστά, τον Γιώχαν Φανόβερφαλτ Βέλπαρτ αντικαθιστά τον κύριο Ραντούτκο και Ρούς αντικαθιστά τον κύριο Βίτο. Για την Γκουε η κυρία Όμπρε αντικαθιστά τον Μάρτιν Σρέντεβαν και η κυρία Μούμερα αντικαθιστά τον κύριο Λόγβερς. Ο κύριος Ντάφνε αντικαθιστά τον κύριο Χάμπιτ και ο κύριος αντικαθιστά τον κύριο Τίς. Υπάρχουν άλλες αντικαταστάσεις, υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη που έχουν πάρει τη θέση κάποιου πλήρους μέλους τακτικού. Όχι, ωραία. Λοιπόν, η απαρτία τώρα για να ισχύσει η ψηφοφορία μας σήμερα έχει επιτευχθεί. 15 μέλη πρέπει να έχουμε, που είναι το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής μας. Υποψηφιότητες τώρα για την εκλογή του Προέδρου. Ο ορισμός μπορεί να γίνει από μία πολιτική ομάδα ή από τρία μέλη. Υπάρχουν υποψηφιότητες, παρακαλώ. Κύριε Ντέλκα. Πρέπει να πάρετε το άλλο μικρόφωνο, Εκ μέρους των σοσιαλιστών θέλω να προτείνω τον κύριο Ρομπέρτο Κολτιέρη ως πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλκα, λέει ο πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλη υποψηφιότητα. Ο υποψήφιος συμφωνεί. Ναι, συμφωνώ, λέει ο κύριος Κολτιέρη. Ευχαριστούμε. Οπότε σημειώνω ότι είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Εκών υποψήφιος και επίσης έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφορώντων του, όπως επίσης και τον κώδικα δεντολογίας. Μπορούμε λοιπόν διαβοής να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα αυτή, εκτός αν κάποιος ζητάει, κάποιο μέλος της ΕΚΟΝ δηλαδή, ζητάει μυστική ψηφοφορία. Το ζητάει κανείς? Αν όχι, ευχαριστώ πολύ και ορίζεται διαβοής εκλέγεται ο κύριος Γκουαλτιέρη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Συγχαρητήρια κύριε Γκουαλτιέρη και εγώ τελείωσα εδώ. Dear colleagues, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι που με εμπιστευτήκατε. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλάβω τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής αυτής. Και δεσμεύομαι να συνεργαστώ μαζί με όλους σας προκειμένου να φέρουμε σε πέρας όσο γίνεται καλύτερα τα καθήκοντά μας. Τώρα θα προβούμε στην ψηφοφορία του πρώτου Αντιπροέδρου. Υπενθυμίζω στους Ευρωβουλευτές επίσης το τι λέει το άρθρο 213.1 που λέει ότι πρέπει η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου μας να αντικατοπτρίζεται στο Προεδρείο, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε Προεδρείο που να αποτελείται από άτομα μόνο του ενός φίλου, ούτε από μία μόνο πολιτική κατεύθυνση. Λοιπόν, υποψηφιότητες. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Παρακαλώ, κύριε Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ Πρώτα απ' όλα σας συγχαίρω για την επανεκλογή σας. Είσαστε από τους λίγους που συνεχίζουν με το αξίωμά του στη θητεία αυτή. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και πάλι στην Προεδρία και ελπίζουμε να έχουμε εξίσου καλή συνεργασία όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Εκ μέρους του ΕΛΚ λοιπόν προτείνω την υποψηφιότητα του κ. Νίτεμάγερ. Συμφωνεί ο υποψήφιος? Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Σημειώνω ότι είναι πλήρε μέλο της επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υποψήφιο και ότι έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση που έχει να κάνει με την διοντολογία. Αν δεν ζητάει κανείς μυστική ψηφοφορία, παρακαλώ διαβοής να κλέξουμε τον υποψήφιο. Uh, Περνάμε τώρα στην δεύτερη αντιπροεδρία. Υπάρχουν υποψηφιότητες παρακαλώ. Ναι, εσείς πρώτα. Κούνο Μπέκ ονομάζομαι και είμαι προσωρινά συντονιστής εκ μέρους της ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας και προτείνω τον κύριο Ρινάλντι, τον συναδελφό μου, για την θέση της δεύτερης αντιπροεδρίας. Κάποιος άλλος έχει ζητήσει όμως να προτείνει υποψηφιότητα. Ναι, εκ μέρου τη ομάδα Renew, Ανανέωση Ευρώπη, προτείνω την συνάδελφο Στέφανη Γιούγκομαλτ. Ωραία, έχουμε δύο υποψηφίου. Δέχονται υποψήφοι. Παρακαλώ. Κύριε Ρινάλντι, εσείς πρώτα. Δέχεστε. Ναι. Ωραία. Τώρα, η δεύτερη υποψήφια. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο Πρόεδρος, έχουμε δύο υποψηφίου για την ίδια θέση. Σημειώνω, λοιπόν, καταρχήν ότι και οι δύο είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και επίσης Διακόπτει ο πρόεδρος. και επίση ότι έχουν και δύο συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών του συμφερόντων και την δήλωση σχετικά με την δεντολογία. Συνεπώ, με μυστική ψηφοφορία ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. για τους υποψηφίους αυτούς. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω, έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, για να κάνουμε μια δοκιμή. Σβέν. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ο κύριος Φίλι Λάμπρεκτς, που είναι τακτικό μέλος, μπορεί να τα κατασταθεί από τον κύριο Καρέμ, που είναι αναπληρωτής στην Επιτροπή αυτή. Καλώς. Η διαδικασία έχει ως εξή. Το πράσινο κουμπί είναι για τον κύριο Ρινάλντι. Πράσινο κουμπί, κύριος Ρινάλντι. Και το άλλο κουμπί είναι για την κυρία Γιον Κουρτέν. Για τις αποχές, το άσπρο που είναι στη μέση, το άσπρο κουμπί. Επαναλαμβάνω, πράσινο κουμπί είναι για τον κύριο Ρινάλντι. Το κόκκινο κουμπί είναι για την κυρία Γιον Κουρτέν. Συμφωνεί. Ας κάνουμε μία δοκιμή πρώτα, όπως κάνουμε πάντα πριν αρχίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία λοιπόν δοκιμαστική έτσι για να ελέγξουμε το μηχάνημα. Είναι μυστική. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Μια στιγμή, μια στιγμή. Πρόκειται για αντικατάσταση. Α. κυρία Άμπραμ θα αντικαταστήσει πρόεδρο. Ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα κανονική ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω, πράσινο κουμπί για τον κύριο Ρινάλντι, κόκκινο κουμπί για την κυρία Γιον Κουρτέν. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Η κυρία Γιον Κουρτέν εκλέγεται με 41 ψήφους. 17 ψήφους πήρε ο κύριος Ζινάλντι. Συγχαρητήρια. Και τώρα Θα εκλέξουμε τώρα ε, τρίτο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Ρόμπερτ Τζίλερ από το ECR. Ήμουν πραγματικό μέλος, τώρα είμαι πλήρως μέλος της Επιτροπής, τακτικό. Εκ μέρους του ECR προτείνω τον Ντέρκεν Έπινγκ σαν υποψήφιο για θέση τρίτου αντιπροέδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο υποψήφιος συμφωνεί με την υποψηφιότητά του. Τη δέχεται, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Σημειώνω που το ψήφιο είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής της Οικονομικής. Επίσης, έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση σχετικά με τα δεντολογικά. Αν δεν απαιτείται μυστική ψηφοφορία, θα γίνει εκλογή διαβοής. Congratulations. Συγχαρητήρια λοιπόν. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο Προεδρείο. Κύριε Πεντιτσίνη. Πρόεδρε, να πω μια κουβέντα. Ήδη στην προηγούμενη θητεία είχα παραστεί σε αυτές τις στιγμές. Εκεί θα έπρεπε να σεβόμαστε μια συμφωνία κυρίων. Έτσι δεν είναι. Όμως όπως και την άλλη φορά χρησιμοποίησατε αντιδημοκρατικές μεθόδους. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα βοηθήσει στο ισορροπημένο κλίμα που θα έπρεπε να επικρατεί κατά τη διάρκεια αυστητία σε αυτή την Επιτροπή. Συνεπώ, εάν όν γίνεται όλοι συνένοχοι, εκείνοι που ψήφισαν τουλάχιστον, σε αυτή τη διαδικασία που είναι αντιδημοκρατική, μη ψηφίζοντα ε, εκείνον που έχει πάρα πολύ διάσημο πρόσωπο, που έχει πολύ σημαντικέ γνώσει για την οικονομία και θα μπορούσε να βοηθήσει όλου μα, τότε θα είσαστε υπεύθυνοι για το γεγονό ότι δεν θα υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα σε αυτή την επιτροπή για όλη τη διάρκεια τη θητεία. Ευχαριστώ, συνάδελφε Πεντιτσίνη. Θα εκλέξουμε τώρα τον τέταρτο ή την τέταρτη αντιπρόεδρο. Υπάρχει υποψηφιότητα. Ορίστε, έχετε το λόγο. Γεια σας. Μανώνο Ομπρί, συντονίστρια για την ομάδα Γκουε και με μεγάλη μου χαρά προτείνω τον Σοζέ Γκουσμάου τον συνάδελφο από την Πορτογαλία για τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου. Ευχαριστώ. Υποψήφιος συμφωνεί με αυτή την υποψηφιότητα. Μάλιστα, Πρόεδρε, συμφωνώ. Σημειώνεται ότι υποψήφιος είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και έχει συμπληρώσει δεόντω ε, τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση σχετικά με τα δεντολογικά ζητήματα. Οπότε διαβοής ας προχωρήσουμε. Ορίστε. Δεν συμφωνούμε με τη μέθοδο διαβοής. Διότι όπως και ο συναδελφός μου είπε ο κ. Πετιτζίνη, ε, και προσπάθησε να κρατήσει την ID από την Επιτροπή και δεν συμφωνώ με την μέθοδο διαβοής και ζητούμε μυστική ψηφοφορία. Ο Jake Pew από το κόμμα Brexit. Δεν έχετε το απαραίτητο όριο των 12 μελών. Δεν έχουμε το απαραίτητο όριο των 12 μελών που μπορούν να ζητήσουν την ψηφοφορία, τη μυστική. Ευχαριστώ. Το όριο δεν επετεύχθη, άρα διαβοής γίνεται η εκλογή. you join? Μπορείτε να έρθετε στη θέση σας εδώ στο Προεδρείο. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη ότι υπάρχουν πακέτα υποδοχής για τα μέλη και βρίσκονται στηρίδες των ε, τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής ΕΚΟΝ και στα επίσημα πακέτα, στο διαδίκτυο επίσης υπάρχουν τα έντυπα, θα βρείτε στο πακέτο αυτό υποδοχή πολλές πληροφορίες για τις διαδικασίες λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο και το πώς υιοθετούνται τα διάφορα νομοθετήματα. Επίσης, συγκεκριμένο βιβλιαράκι που ετοίμασε η Γραμματεία για την οικον και πληροφορίες για τις διάφορε ε, ε, διάφορες υπηρεσίες που διατίθενται στα μέλη για το κοινοβουλευτικό του έργο. Να πω σε όλα τα μέλη επίση ότι λάβαμε αποφάσεις σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπανε την εκλογή προέδρων και την προέδρων. Σεβαστήκαμε τους κανονισμούς. Καλό τα μέλη να συμβάλλουν στις εργασίες, να υπάρξει πλήρης συνεργασία. Να τιμήσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε το έργο μας που είναι πολύ ευαίσθητο και σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλές ευθύνες αυτή την Επιτροπή, οικονομικού είδους αλλά και για θέματα πολιτικού ελέγχου της Τραπεζικής Ανώσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα έχουμε σημαντικότατα καθήκοντα να εκτελέσουμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και ξανά επαναλαμβάνω ότι είμαστε, είμαι αφοσιωμένος να συνεργαστούμε ε, με όλα τα μέλη της Επιτροπής. Συνεργαστώ με τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τις συνεδρίες. Έχετε πρόγραμμα ημερήσια διάταξη προσωρινή για την επόμενη συνεδρίαση. Θα κάνουμε έναν έλεγχο με τη γραμματεία να δούμε κατά πόσο είναι σωστά αυτά τα σημεία. Περιμένετε μία-δύο ώρε, ούτω ώστε να λάβετε το τελικό έγγραφο, τελική ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση. Πότε θα γίνει και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδριά σου.